Παρακαλώ καθίστε. La séance ouverte. Ξεκινάει η συνεδρίαση. Οι διερμηνείς ε, έχουν μια δήλωση να κάνουν. Μας είπαν ότι η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώς στις 10.30 θα είναι πολύ αυστηρή με το ωράριο, οπότε θα είμαστε και εμεί αυστηροί με την ε, εξέτηση τη ημερήσια διάταξη. Βρισκόμαστε στην 24η μέρα των κινητοποιήσεων ε, των διερμηνέων λόγω της ε, δυσκολίας συνεννόησης με τη Γενική Γραμματεία. Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι η διερμηνία θα διακοπεί ακριβώ στι 10.30. Λοιπόν, θα θεωρήσουμε ότι η μερίσια διάταξη έχει εγκριθεί, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, Διευκρινίζω ότι θα γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση Badge Econ 2 Ιουλίου στο Στρασβούργο για το Invest EU. Για το Invest EU. Βλέπω τώρα ότι η μελέτη που ζητήθηκε από το θεματικό τμήμα η για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ε, παράτασης του συστήματος ε, χρηματοδότησης ε, μέσω τελών ορισμένων οργανισμών μετά από μια διαδικασία αποστολής προσφορών δόθηκε η εντολή ε, για τη διεξαγωγή αυτή τη μελέτη. Ε, από το γραφείο Deloitte έχουν έρθει σήμερα εδώ για να μας δείξουν τα αποτελέσματα της έρευνας ε, αυτής. Οι κύριοι Βαν Σχόμπροκ, Σονιέ και Λενό. Χωρίς άλλη καθυστέρηση δίνω το λόγο στον εισηγητή μας, κύριο Γκάιερ, για μια σύντομη εισαγωγή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η χρηματοδότηση των οργανισμών αυτών ε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ε, αρκετό καιρό τώρα. Η κατάσταση υπήρξε κάπως κρίσιμη όσον αφορά τα έσοδα των οργανισμών αυτών. Ο οργανισμός του Αλεκάντε έχει προβλήματα όσον αφορά τα τέλη και την αφάνεια των κανόνων, το γεγονό ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα με άλλου τρόπου. Υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που δεν προσφέρουν καν ε, υπηρεσίε που βάσει των οποίων μπορούν να ζητήσουν ε, τέλειο ώστε να επαναχρηματοδοτήσουν ε, το, αυτούς τους ο προπολογισμό του είναι σχετικά μικρό σε σχέση με το συνολικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αν είναι να μιλάμε για γενικές οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο που σκέφτεται κανεί είναι οι οργανισμοί, διότι είναι τόσο πολλοί και κανείς δεν έχει μια σαφή εικόνα του τι ακριβώς κάνουν. Γι' αυτό το λόγο, ω εισηγητή για του ε, οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ήθελα να προσπαθήσω να απαλύνω κάπω την πίεση προσπαθώντας να βρω τρόπους να προχωρήσουμε μαζί με τους οργανισμούς, να δούμε πώς μπορούμε λοιπόν να μειώσουμε ουσιαστικά τη συμμετοχή από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό στους οργανισμούς αυτούς και να βρούμε άλλες πηγές χρηματοδότησης για τους οργανισμούς αυτούς. Χαίρομαι που η Επιτροπή αποφάσισε να ε, ζητήσει μια σε βάθος ε, μελέτη και το ανέθεσε στην Deloitte. εταιρεία που μας έχει δείξει ήδη την εμπειρογνώμοσύνη της επί του θέματος σε διάφορες ευκαιρίες. Οπότε έχουν έρθει εδώ σήμερα για να μας δείξουν τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε κύριε εισηγητή. Το λόγο έχουν οι εμπειρογνωμονές μας. Ο κύριος Τιέρι Βαν Σχόμπροκ ε, να μας παρουσιάσει τη μελέτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γκέρ, για την ε, εισαγωγή που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα της μελέτης μας εδώ σήμερα. Να σας υπενθυμίσω ότι πεδίο αντικείμενο της ε, μελέτης μας ήταν 33 αποκεντρωμένοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έσοδα άνω των 3 δισεκατομμυρίων, με προπολογισμό άνω των 3 δισεκατομμυρίων για το 2018 ε, εξετάσαμε το πιθανά έσοδα, το τι θα γίνει στο μέλλον, τα πιθανά Οφέλη και τα συμπεράσματά μας ε, βασίζονται στην αναθεώρηση σε πολλές συνεντεύξεις με τους ενδιαφερομένους, με τους θεσμικούς ενδιαφερομένους. Πραγματοποιήσαμε και μια έρευνα που έγινε στους περισσότερους οργανισμούς, 24 από τους 33 ε, και σε βάθος συζητήσει με έξι οργανισμούς ΆΣΕΡ, ΕΑΖΑ, ΕΡΑ, ΕΦΣΑ, ΕΣΜΑ και ΕΚΑ που εκπροσωπούν την ενέργεια, την αεροπλοεία, τα χημικά, την ασφάλεια και τις αγορές. Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάσαμε δύο τύπους δραστηριοτήτων. Πρώτον, εξουσιοδότησης, πιστοποίησης, έγκρισης, ε, καταχώρησης και εξαίρεσης όπου μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε έσοδα. 34% ουσιαστικά των εσόδων ε, λίγο παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο ε, ε, αντιπροσωπούν, εκπροσωπεύουν αυτά τα έσοδα. Εξετάσαμε τις δυνατότητες εξωτερικής χρηματοδότησης αυτών των οργανισμών. Στο πλαίσιο των εποπτικών δραστηριοτήτων αντιληφθήκαμε ότι υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες δημιουργίας τέτοιων εσόδων. Ουσιαστικά Έχουμε και η WIPO, SRB που είναι πλήρως χρηματοδοτούμενε, αυτοχρηματοδοτούμενες και μετά συγχρηματοδοτούμενου οργανισμούς έχουμε την ΕΑΣΑ 60 έως το 80% ε, αυτοχρηματοδοτείται ανάλογα με το έτος. Η ΕΚΑ 40 έως 80% και η ΕΣΜΑ περίπου 26%. Οι οργανισμοί χωρί εποπτικές δραστηριότητε δεν έχουν τέτοια έσοδα. Και μετά έχουμε το δεύτερο τύπο δραστηριοτήτων. Αυτό αναφέρεται ως χρεώσεις για υπηρεσίες που παρέχονται και πληρωμές ε, έναντι υπηρεσιών. Έχουμε διάφορε δραστηριότητε, δημοσιεύσει, εκπαίδευση, επεξεργασία δεδομένων, έρευνε, συντονισμό κτλ. 19 οργανισμοί τέτοιοι προβλέπουν ότι έχουν τη δυνατότητα τώρα να χρεώνουν εξωτερικού ενδιαφορουμένου για οποιασδήποτε υπηρεσίε παρέχουν τέτοιου είδου. Αλλά σήμερα μόνο τέσσερι από αυτού ε, εφαρμόζουν τέτοιου είδου ε, χρηματοδότηση. Εδώ μιλάμε για τον CDFOP, EASA, EMA και Eurofound. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι δραστηριότητε αυτέ δημιουργούν αυτή τη στιγμή το 0,02% του συνολικού προπολογισμού των οργανισμών αυτών, λιγότερο από ένα εκατομμύριο δηλαδή. Οι δυνατότητε περαιτέρω επέκταση τέτοιου είδου χρηματοδότηση είναι περιορισμένε, διότι πρώτα απ' όλα σε πολλέ περιπτώσει ο τύπο ε, δραστηριοτήτων στον οποίο αναφερόμαστε θεωρούνται δημόσια αγαθά ή δημόσιε υπηρεσίε, οπότε πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Και επίση ο, ο όγκο των δραστηριοτήτων, των δραστηριοτήτων αυτών είναι περιορισμένο σχετικά. Οπότε η εσωτερική χρηματοδότηση δεν είναι ικανοποιητική. Σχετίζεται με μικρά ποσά, αλλά και ποσά τα οποία δεν είναι πολύ προβλέψιμα ούτε σταθερά από τη φύση τους. κάποια μαθήματα που έχουμε αποκομίσει από την έρευνα αυτή είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι πρωτοβουλίε για λιγότερη πίεση στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, για αύξηση των προπολογισμών των οργανισμών ε, είναι ευπρόσδεκτε από όλου του ενδιαφερομένου. Ε, οι πρωτοβουλίε αυτέ μπορεί να σχετίζονται με αύξηση των τελών και με άλλε πηγέ ε, χρηματοδότηση, χορηγίε, συμβολέ από τρίτε χώρε μέσα στα επόμενα χρόνια μπορεί να εξεταστούν και αυτά τα ενδεχόμενα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα έσοδα των οργανισμών θα χρηματοδοτούνται ως επιτοπλίστων ε, και στο μέλλον από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Αυτή τη στιγμή ο οικονομικός κανονισμός, ο δημοσιονομικός κανονισμός δεν αλλάζει προσέγγιση για τη χρηματοδότηση των οργανισμών. Ορισμένοι χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, η Άσερ και η ΕΦΣΑ για παράδειγμα παρότι έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίε ε, χρηματοδότησης μέσω τελών, αλλά απέχουμε πολύ από τον τελικό σχεδιασμό ή την υιοθέτηση του ε, σχετικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για να είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Επίσης ξέρουμε ότι η επέκταση της ε, διαδικασίας τελών είναι περιορισμένη. Αυτό το είδαμε και στην απαλλαγή του Κοινοβουλίου του 2015 για τη ΣΕΦΣΑ και την ΕΜΑ. Υπάρχουν κάποια ωφέλη όσον αφορά τα συστήματα τελών, αλλά και κάποιοι περιορισμοί. Όσον αφορά τα ωφέλη από επιχειρησιακή και δημοσιονομική οπτική γωνία, τα τέλη φέρνουν τους οργανισμούς πιο κοντά στην αγορά, βοηθούν στην βελτίωση του σχεδιασμού, καλύτερη απόκριση στις ανάγκες των ενδιαφερομένων, καλύτερη εκτέλεση του προπολογισμού, ε, πιο ακριβής ε, κατανομή των πόρων και πιο αποτελεσματική. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί και από άποψη προσωπικού και δημοσιονομική. Η χρηματοδότηση μέσω τελών δεν παρέχει καλύτερη ευελιξία στα σχέδια ε, σύστασης και δεν σημαίνει αυτό ότι οι προπολογισμοί αυξάνονται εκ των πραγμάτων. Όποιο μοντέλο τελών και αν υιοθετηθεί, η εμπειρία δείχνει ότι είναι σημαντικό να δοθεί επαρκής προσοχή στην αντιστάθμιση μεταξύ διαφάνειας και πολυπλοκότητας ε, διαχείρισης των ε, τελών. Τα κόστη πληροφορικής, ε, τα διαχειριστικά κόστη μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία για το σχεδιασμό ενός μοντέλου τελών. Σε αυτό το πλαίσιο τόσο η Κομισιόν όσο και η Δημοσιονομική Αρχή υποστηρίζουν απλούς μηχανισμούς υλοποίησης ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη που θα προκύψουν από την εισαγωγή των συστημάτων τελών. Going into a little bit of the details, uh, generally agencies would... Μπαίνοντα σε λεπτομέρειε, σε ό,τι αφορά τι δραστηριότητε καταχώρηση, εδώ υπάρχει ένα δυναμικό χρηματοδότηση μεγαλύτερου τμήματο ε, των τελών, αλλά η αύξηση τη χρηματοδότηση ε, με βάση τα τέλη δεν θα υπερβεί το 3% κατά Δηλαδή το 34% που έχουμε σήμερα μπορεί να φτάσει στο 37% ενδεχομένω βάσει ε, ορισμένων πρωτοβουλειών. Το γράφημα που βλέπετε εδώ περιγράφει το πιθανό μέλλον για την χρηματοδότηση από τον κλάδο. Στον άξονα Χ βλέπετε το πιθανό ποσοστό επιλέξιμων δραστηριοτήτων για έναν οργανισμό, ενώ ο άξονα Ψ εστιάζει σε στοιχεία που συνδέονται με την εφικτότητα των δραστηριοτήτων αυτών, δηλαδή πολιτική βούληση, ύπαρξη νομικής βάσης, ε, πρόοδο στην διαδικασία της επιτροπολογίας, αποδοχή του κλάδου, κόστος εφαρμογής και το καθεξής. Από το μέγεθος του κάθε κύκλου βλέπετε τις δυνατότητες που έχουν, έχει ο κάθε φορέας. Οι πράσινες πισαλίδες που βλέπετε στο γράφημα παραπέμπουν σε οργανισμούς όπου υπάρχει status quo ε, ρύθμισης τελών, όπου δεν αναμένεται κάτι παραπάνω. Αν χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της ε, ΕΚΑ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προγραμματισμένη πρωτοβουλία για την εισαγωγή νέων ε, δραστηριοτήτων χρηματοδότησης για τον ECA. Όμως τα τέλη, τα ιδιωτικά τέλη του κλάδου δηλαδή, ε, αναμένεται να μειωθούν κατά το ίμιση σε σχέση με τα βίδα του 18. Δηλαδή η συνολική προγραμματισμένη αύξηση του 3% αντισταθμίζει την αναμενόμενη μείωση του ECA με αύξηση ε, στις δυνατότητες που έχουν άλλοι οργανισμοί. Αυτά έχουμε βάλει ε, σε μπλε χρώμα. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες ευρωπαϊκές αρχές που μπορούν να παρατείνουν ή να επεκτείνουν ε, τις ε, χρεώσεις και τη χρηματοδότηση μέσω χρεώσεων. Η ΆΖΑ ε, που μπορεί να ρυθμίσει τα drones, εισαγωγή πιθανής επιπρόσθετης χρηματοδότησης στην ERA με το τέταρτο συνδρομικό πακέτο για τον ΕΜΠΑ, ΕΟΠΑ και ΕΣΜΑ. Το θέμα είναι να από τα, τις χρηματοδότητες με τα κράτη-μέλη να περάσουμε σε τέλη από τον κλάδο. Εξετάζουν οι οργανισμοί αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο επιβολή ε, τέτοιων τελών. Για παράδειγμα, ο Acer έχουν προσθεκοποιήσει δραστηριότητε που μπορούν να οδηγήσουν σε χρηματοδότηση ε, σημαντική για ένα συνολικό προπολογισμό 9-10 εκατομμυρίων. Και η ΕΦΣΑ εξετάζει πιθανή ανασκόπηση για μηχανισμούς ε, χρηματοδότησης σε δραστηριότητες όπως ε, η παροχή υπηρεσιών σε ετούντες, παρακολούθηση ε, δραστηριοτήτων και το καθεξής. Ήδη υπήρχε πρωτοβουλία το 2012, μια μελέτη αντικτύπου για τα τέλη και τότε δεν είχε δοθεί το πράσινο φως για την επιβολή τελών από την ΕΦΣΑ. Τέλος, για την ΕΜΖΑ. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι καλό θα ήταν και ότι είναι κατάλληλοι για να τις ε, εμπιστευτούμε τέτοιου είδου δραστηριότητε. Τώρα είναι πολιτική απόφαση από εκεί και πέρα. Οι υπόλοιποι 21 ε, φορεί που εξετάσαμε δεν ε, είδαν τέτοιες δυνατότητες για υπηρεσίες με βάση τα τέλη. Η πιθανή αύξηση αυτής της χρηματοδότησης θα αποτελέσει τμήμα του επόμενου ΠΔΠ. Ακόμα Υπάρχει μια αμφισημία σε ό,τι αφορά το, τους έμεσους δικαιούχους που συνδέονται με τον ΕΜΠΑ, τον ΕΟΠΑ και, το, και την ΕΣΜΑ και υπάρχει μια πρόταση να ξεμπλοκαριστεί αυτό το πρόβλημα ε, που αναμένεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβρη. Πέραν τούτου, ανέφερε και προηγουμένω τα διάφορα επίπεδα προόδου, πρωτοβουλίε ε, για την υλοποίηση των, του συστήματος επιβολής ε, τελών, όπω βλέπετε και στο επόμενο γράφημα. Η ΕΦΣΑ και ο ΕΙΣΕΡ βρίσκονται στα προκατακτικά στάδια στην ίδια τους ε, την ύπαρξη, ενώ οι υπόλοιποι πέντε οργανισμοί είναι στη διαδικασία επιτροπολογίας αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι φορά τα συμπεράσματα, οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που έχουν δραστηριότητε επιλέξιμε για τέτοια χρηματοδότηση ήδη συλλέγουν τέλη σήμερα ανέφερα το 34% του προπολογισμού των ε, οργανισμών αυτών που ανέρχεται στο 1 δις. Το ποσοστό των ε, δραστηριοτήτων αυτών που είναι επιλέξιμες ε, τελών δεν αναμένεται να αυξηθούν. Υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες που είναι επιλέξιμες για τέτοια χρηματοδότηση και πολλές πρωτοβουλίες είναι καθοδόν. Ε, το γεγονός ότι δεν είναι πολλέ αυτές οι δυνατότητε δεν ε, προβληματίζει ιδιαίτερα πολλά ενδιαφέροντα μέλη. Ε, οι οργανισμοί θα ενημερώνονται και τις δραστηριότητε τους με ικανοποιητικό τρόπο και με βάση τις σημερινέ και μελλοντικέ δυνατότητες χρηματοδότηση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να υπάρχουν δραστηριότητες που είναι επιλέξιμε για χρεώσει τελών και δεν χρεώνουν, αναφέραμε ορισμένε, υπάρχει δυνατότητα να διαρευνήσουν αυτές τις ευκαιρίες, λαμβάνοντα υπόψη ότι ε, συνήθως τα ωφέλη τέτοιων συστημάτων αντισταθμίζουν και είναι περισσότερα ουσιαστικά από τα μειονεκτήματα. Αν δημιουργηθούν νέοι οργανισμοί ή αποφασίσουν Καλό είναι να αποφασίσουν από την αρχή αν θα επιβάλλουν ένα τέτοιο σύστημα επιβολή τελών για λόγους εναρμόνισης ε, και με τις ε, ευρωπαϊκές πολιτικές ε, η επιβολή από την αρχή αυτών των συστημάτων μπορεί να μειώσει το διοικητικό άχθος. Τέλος. Θα πρέπει να αποφύγουμε ένα υπερβολικά σύνθετο σύστημα κατά το δυνατόν. Κλείνω εδώ τα εισαγωγικά μου σχόλια και με τα χαράς να ακούσω τα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Στρέφομαι στον εισηγητή, τον μόνιμο εισηγητή, Γιάννης Γκάιερ. Μήπως έχετε κάποιες πρώτες παρατηρήσεις? Äh, Ευχαριστώ και έχω και θα πω τις παρατηρήσεις μου. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά στη μελέτη για τα οποία με τις εργασίες της Επιτροπής μας θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια επιρροή για να δώσουμε μια καθοδήγηση ως προς την ποια κατεύθυνση θα πρέπει να οδηγηθούμε με την επέκταση αυτή των τελών για ορισμένους εκτελεστικούς οργανισμούς και νομίζω ότι ως προς αυτό ήταν καλή μελέτη, αλλά είμαι και κάπως απογοητευμένος. 37% λέτε είναι το μέγιστο ποσοστό, θα ήθελα λίγο παραπάνω. Αλλά αν έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά βλέπω ότι υπάρχει ένα δυναμικό δυνατό τις οποίες σχεδόν τις έχουμε εξαντλήσει. Μιλήσατε για κάποιους δύο οργανισμούς που μπορούμε να έχουμε κάποιες θετικές και στο μέλλον. Επίσης, στις συζητήσεις που θα έχουμε εμείς, όλα αυτά που είπατε θα παίξουν το ρόλο τους. η δεξιά πτέρυγα στο κοινοβούλιο ανησυχεί ε, με αυτή τη θέσπιση τελών, ότι μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη επιβάρυνση της οικονομίας. Τελικά βλέπουμε όμως ότι και πιο κοντά στην αγορά έρχονται και καλύτερο σχεδισμό μπορούν να κάνουν ε, και να καλύψουν περισσότερες ανάγκες των εμπλεκομένων. Επομένως φαίνεται να μην είναι τόσο άσχημο κάτι τέτοιο ως προοπτική. Χρειάζεται βέβαια ε, μια ε, εντατικοποίηση της συνεργασίας των φορέων της αγοράς και των ε, οργανισμών. Δεν ξέρω αν μπορείτε κι εσείς ε, να μας δώσετε περισσότερα ε, στοιχεία με κάποια παραδείγματα ενδεχομένως. Ε, οι συνάδελφοι λοιπόν από τη δεξιά πατέρυγα χριστιανοδημοκράτες, φιλελεύθεροι έχουν τα δικά τους μάτρα και τα δικά τους σλόγγαν, αλλά νομίζω ότι αυτά που βλέπουμε, τα πορίσματα αυτής της μελέτης της Deloitte, δείχνει ότι είναι θετικό αυτό το μέτρο για τους οργανισμούς και αυτό είναι βοηθητικό. Υπάρχει μια ένσταση βέβαια σε ό,τι αφορά ε, την ε, αμφισβήτηση της αυτονομίας ενδεχομένως ε, και ανεξαρτησίας αυτών των οργανισμών με την αύξηση των τελών. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχήσουμε σοβαρά, αλλά θα ήθελα να μας δώσετε κι εσείς να μας καθιστικάσετε δίνοντάς μας κάποια παραδείγματα από αυτού. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι προκλήθηκαν κάποιες αντιδράσεις, ε, κύριε Μόνιμη Σιγητά, από κάποια από τα σχόλιά σας. Δεν κατάλαβα κάτι πολύ καλά με, αυτή την, ε, με αυτά τα τέλη και, και την ε, ανεξαρτησία οι φορολογούμενοι που πληρώνουν ε, φόρους ε, χάνουν την εξαρτησία τους. Ε, δεν έχω πολύ καλά καταλάβει αν υπάρχει ρύθμιση, νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται σε όλους. Και αυτό το 37% και εγώ δεν το κατάλαβα. Να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Η κυρία Γκρέσλε. Το μάτρα μας ε, δεν είναι αυτό που είπατε εσείς. Ε, ε πάντων, έχω κάποιες ερωτήσεις. Δεν ε, κατάλαβα πολύ καλά τι γίνεται σε σχέση με το δημοσιονομικό κανονισμό αυτών των οργανισμών. Δεν θα ισχύει πλέον το οργανόγραμμα, δεν θα ισχύει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Αυτό θα είναι πρόβλημα, γιατί ήταν μια εγγύηση για να μην υπάρχουν υπερβολές μέχρι τώρα. Αλλιώ θα υπήρχαν υπερβολέ. Ε, είμαι πεπισμένη. Λόγω τη κεντρική αυτή διαχείριση των οργανισμών. Και στην απαλλαγή έχουμε τη δυνατότητα έτσι ε, να δούμε πράγματα που ίσως ως βουλευτές δεν θα μπορούσαμε να δούμε, δεν θα είχαμε πρόσβαση. Και σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα αυτών των τελών, δεν έχω διαβάσει τη μελέτη, ελπίζω να τα καταφέρω σύντομα. αλλά έχω δει για ε, κάποιον οργανισμό, την ΕΚΑ συγκεκριμένα, να γίνει ε, μεγάλος χαμός από τις επιχειρήσεις με ένα μεγάλο ποσοστό. Άρα, ναι μεν μπορεί να λειτουργήσει το ποσοστό, αλλά ε, θα πρέπει να αποφευθούν επιθέσεις έξωθεν. Και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τους μεγάλους και τους μικρούς. Οι μεγάλοι ε, σίγουρα θέλουν να διώξουν τους μικρούς από την αγορά με τη βοήθεια αυτών των τελών. Τι διασφαλίσεις υπάρχουν για να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Βλέπουμε τους παπτικούς οργανισμούς, ε, βλέπουμε τους άλλους οργανισμούς. Ε, ε, νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Έχω συμπάθεια προς τους ελεγκτές, αλλά υπάρχει το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σοβαρά. Και θα ήθελα να μας πείτε κάτι από αυτού. Euh, Κύριε Ρούμπιχ, ευχαριστώ. Είναι ένας ενδιαφέρον ε, τομέας αυτός ε, για τους οργανισμούς αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που ιστορικά έχουν εξελιχθεί, κίνησαν με κάποιες δομές, κάποια καθήκοντα και εξελίσσονται. Το ερώτημα είναι αν να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα και τα καθήκοντα των οργανισμών. Ήδη αυτοί οι οργανισμοί είναι ισχυροί γιατί παράγουν πολλή γνώση. Ε, και νομίζω ότι από αυτούς τους οργανισμούς προκύπτει μεγάλη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Ένα ερώτημα είναι πώς μπορούν να τους διαδικτυώσουμε μεταξύ τους καλύτερα αυτούς τους οργανισμούς. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει μία εναρμόνιση ε, κάποιας ε, επιχειρησιακής βάσης αυτών των οργανισμών μπορούμε να το σκεφτούμε. Και βέβαια η επικοινωνία είναι ένα άλλο θέμα, η επικοινωνία μεταξύ των οργανισμών. Από τους 44 οργανισμούς νομίζω ε, πάνω από 400 οργανισμοί, ε, ε, υπάλληλοι πάνω χάρη σε έναν οργανισμό. Ε, ρωτήσαμε πόσους ξέρετε, ποιες άλλους, ποιους άλλους οργανισμούς ξέρετε και ήταν πάρα πολύ λίγο το ο αριθμός, 5, 10... Ε, εντάξει, ήταν ως αστείο, αλλά πραγματικά υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει ε, μια κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών. Ίσως θα πρέπει να διαρθρωθεί αυτή η συνεργασία, να είναι προσανατολισμένη προς τους στόχους δε αυτή η συνεργασία. Έσα, Μπέρεκ, Ενίζα είναι παραδείγματα. Αν θέλουμε να έχουμε μια ψηφιακή αγορά, με εφή δίκτυα και τα δίκτυα παροχής ε, φυσικού αερίου θα πρέπει να συνεργάζονται ως προς αυτούς τους σκοπούς αυτοί οι τρεις οργανισμοί. Δεν υπάρχει δομή όμως ως προς τη συνεργασία ή ως προς την επικοινωνία μεταξύ αυτών των οργανισμών. Και επίσης δεν έχει αξιολογηθεί και το πώς ε, γίνεται αυτή η επικοινωνία και νομίζω ότι πρέπει εδώ να αναλάβουμε επιγόντως δράση και να δούμε αφενός ναι με να μην ασκούμε μεγάλη επιρροή στους οργανισμούς, αλλά να μπορέσουν οι οργανισμοί αυτοί να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά μεταξύ τους. Όσο πιο ε, μεγάλη ο χρήστης, ε, τόσο πιο πολύ φαίνεται και το κόστος από τη μη Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε όλες τις επιπτώσεις αυτής της ε, θέσπισης τελών και να δούμε ε, ποιοι θα ωφεληθούν, περισσότερο πώς μπορούμε να ωφελήσουμε ε, και τους χρήστες, άρα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία, καταρχάς επικοινωνία μεταξύ των οργανισμών, όπως είπα, και φεύγει επικοινωνία με τους χρήστε και πληροφόρησή του. Γιατί πρέπει και οι πολίτε μα να γνωρίζουν τι γίνεται. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω οικονομικά από ιδεολογική άποψη στον συνάδελφο Γκάιερ. Δεν είναι αυτό που θα μας απασχολήσει σήμερα. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει ως εξής. Όταν λέτε ότι το ποσοστό εσόδων μπορεί να περάσει από το 34% στο 37% βασίζεστε σε τι, πού βρίσκεται αυτή η αξιολόγηση, βάσει ποιων παραμέτρων λέτε κάτι τέτοιο, ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε για κάτι παραπάνω. Και αντικειμενικά, τι σημαίνει αυτό υπό απόλυτους όρους. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη μου ερώτηση έχει ως εξής ήθελα να κάνουμε μια σύγκριση με τα εθνικά κράτη όπου έχουμε μια κεντρική φορολογική διοίκηση αρμόδια για την ε, ίσπραξη των διαφόρων φόρων. Εδώ όπως κατάλαβα ο κάθε οργανισμός πρέπει να οργανώσει μόνος του το δικό του σύστημα ίσπραξης ε, τελών, των τελών αυτών από τους υποχρεούς. Έχετε μελετήσει κάτι ή αυτό είναι εκτός κάθε... Δηλαδή ουσιαστικά ρωτάω αυτό που ρώτησε και ο συνάδελφός. Έχετε αποκλείσει το να υπάρχει κάποιο είδους σύστημα κατάρτισης ε, γιατί έχουμε 36 οργανισμούς, έχουμε μια υπηρεσία διαχείρισης προσωπικού, μια υπηρεσία ίσπραξης ε, ε, δημοσιονομική υπηρεσία ουσιαστικά και μια υπηρεσία ίσπραξης των τελών θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο εναλλακτικό σύστημα οικονομικά πιο αποδοτικό όντας παράλληλο εξίσου, παράλληλα εξίσου αποτελεσματικό αλλά κοστίζοντας λιγότερο. Thank you, uh, Mr. President. Uh, Mr. Uh Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντεπρέ. Ρωτήσετε αυτό το παραπάνω 3% τι σημαίνει σε θέματα συνολικής συμβολής στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι που το ακούω ε, για το ιδεολογικό πείραγμα του συναδέλφου. Αναφέρατε για την ανεξαρτησία των οργανισμών και πιθανό συμβιβασμό μέσω της ε, επιβολής τελών. Το επόμενο ιδεολογικό βήμα θα ήταν να πούμε ότι η ρυθμιστική λειτουργία, ε, ο ρυθμιστικός ρόλος των οργανισμών θα μπορούσε να αποβεί εποφελής μέσω της ανάθεσης ε, αυτής της λειτουργίας σε κάποιους ιδιώτες, δημιουργώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο για, τις, ε, για την εκτέλεση των, λειτουργικών, των αριθμιστικών λειτουργιών. Είναι μια έξυπνη ιδέα, αλλά εγώ είμαι κατά, διότι η εμπειρία μας δείχνει ότι δημιουργεί πρόβλημα στη ρυθμιστική λειτουργία. Δεν θα είναι δυνατή η παροχή μια υπηρεσία σωστή λόγω της ανταγωνιστικότητας. Αυτό που προτείνω είναι ότι αν οργανισμοί οποιοδήποτε επίπεδου χρεώνουν ε, κάποιους για να παρέχουν υπηρεσίες, ε, τα τέλη αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από κάποιο σύνολο ε, επίπεδων απόδοσης. Τι είδους υπηρεσία μπορεί να αναμένει κανεί από τον οργανισμό, δηλαδή, αντί να μιλάμε για άλλη μια απομακρυσμένη γραφειοκρατία, στην οποία κανείς πληρώνει τέλη Επίσης να ρωτήσω μέσω εσά, κύριε Πρόεδρε, του εμπειρογνώμονε εδώ, όταν μιλάμε για μια πιθανή, ένα πιθανό νέο τέλος, τι χρόνος αποπληρωμής θα θεωρείτε, γιατί αυτό αποτελεί σημαντική αλλαγή όσον αφορά το κόστος για οποιονδήποτε εμπλέκεται με οποιονδήποτε οργανισμό. Και εδώ τίθεται το θέμα που έθεσε ο κύριος Ντεπρέ τι είδου γραφειοκρατικό πλαίσιο θα έχουμε για αυτούς 30 και παραπάνω οργανισμούς οι οποίοι θα χρεώνουν λογιστικά, γραφειοκρατικά, όλα αυτά πώ θα το ε, κάνουμε να είναι πιο ομαλό. Ευχαριστώ κυρία Τωμά. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois que, en fait... Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. είτε το τέλος θα είναι μία κατά οικονομική συμμετοχή ανεξαρτήτως της υπηρεσίας που παρέχεται αναλογική ως προς τίποτα ουσιαστικά δεν θα είναι αναλογική θα είναι ένα ποσό εφάπαξ σταθερό το οποίο καταβάλλεται για οποιονδήποτε οργανισμό ο οποίος θα σχετίζεται με τις δραστηριότητες του οργανισμού ή θα αγοράζει υπηρεσία στον οργανισμό θα μιλάμε για ένα σταθερό ποσό που σε τελική ανάλυση δεν θα βαρύνει όσον αφορά την επιλογή του οργανισμού. Αντιθέτως, αν μιλάμε για αμοιβή έναντι υπαρχής υπηρεσίας, αναλογική δηλαδή με την υπηρεσία, με το χρόνο εργασίας ε, του οργανισμού και την τεχνογνωσία του οργανισμού, η αναλογική με το μέγεθος επιχείρησης ε, δεν έχει σημασία. Εκεί αλλάζει φύση. Το τέλος αυτό. Και δυστυχώς όπως έχουμε δει κύριε Ντεπρέ, το θέμα εδώ δεν είναι ιδεολογικό. Πολλές φορές ε, για οργανισμούς πολύ ε, υψηλών επιδόσεων έχουμε παρατηρήσει ότι επειδή δεν χρηματοδοτήθηκαν επαρκώ από κοινότητε ή ε, δημόσιους προϋπολογισμούς ε, χρειάστηκε να χρεώσουν ε, τις υπηρεσίες τους και εκεί, και ξαναλέω δεν είναι ιδεολογικό εδώ, είδαμε ότι άλλαξαν οι στόχοι ουσιαστικά των οργανισμών αυτή, αυτών διότι για να χρηματοδοτηθούν τελικά εγκατέλειπαν τις αποστολές γενικού συμφέροντος που δεν ήταν αποδοτικές υπέρ αποστολών, υπέρ δραστηριοτήτων για επιχειρήσεις που αποτελούσαν και την οικονομική τους πηγή. Λέγοντα αυτό, σκέφτομαι διάφορου οργανισμού στη Γαλλία. Ε, συγγνώμη κύριε Τεπρέ, λέω αυτά που γνωρίζω και έχετε φυσικά το δικαίωμα να πείτε κι εσεί αυτά που γνωρίζετε εσεί. Ε, σταδιακά λοιπόν οι οργανισμοί αυτοί, αυτά τα θεσμικά όργανα, άλλαξαν μορφή και δεν επιτελούσαν πλέον ε, κάποιο, κάποια αποστολή ε, δημοσίου συμφέροντο. Το ερώτημα είναι λοιπόν πώ θα συνδυάσουμε την ε, αμοιβή από, από τρίτους που χρησιμοποιούν έμεσα, επωφελούνται κατά κάποιο τρόπο από τις δραστηριότητες, τις επιδόσεις και την τεχνογνωσία των οργανισμών αυτών και πώς θα προστατεύσουμε ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον που από... δεν θέλουμε να εξαφανιστεί υπέρ των ιδιωτικών ε, στόχων οπότε τίθεται ένα ζήτημα περιορισμού εδώ των ε, δραστηριοτήτων και πώς καθορίζουμε το τέλος επίσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα μιλάμε για μία καταποκοπή ε, πληρωμή για μία υπηρεσία ε, ή θα είναι σε ίδιο επίπεδο για όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως ε, υπηρεσίες που παρέχεται. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο από τους συναδέλφους. για να γίνει ακόμη πιο ευανάγνωστη και ευνόητη η έκθεση, καλό θα ήταν να υπάρχει και ένα γλωσσάρι, γιατί κάπου χανόμαστε με όλα αυτά τα αρτικόλεξα. Νομίζω ότι θα μας βοηθούσε να έχουμε κατά νου τον στόχο ε, του κάθε οργανισμού με αυτόν τον τρόπο, το οποίο δεν είναι πάντα ε, ευνόητο με βάση το αρτικόλεξο. Επίσης θα πρέπει να αιτιολογήσουμε γιατί ε, μένουμε στο 37%. Ίσως εδώ ο κύριος Σοερόλη θα μπορούσε να πει ποια είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω αρχικά τον Γενικό Εισηγητή κύριο Γκάιερ και την Επιτροπή σας ε, που ανέλαβε την πρωτοβουλία για αυτή τη μελέτη που μας δίνει μια καλύτερη εικόνα του σύνθετου αυτού ζητήματος. Όπως προτείνεται και στην μελέτη, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της διερεύνησης δυνατοτήτων περαιτέρω χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών οργανισμών με σκοπό να περιοριστεί το άχθος ε, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και έτσι θεωρούμε ότι αυτή η μελέτη ε, είναι σημαντική συμβολή στη συζήτησή μας. Όμως είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε, όπως ανέφερε η κυρία Γκρέσλε, ότι πρέπει να υπάρξουν και κατάλληλες διευθετήσεις ε, χρηστής διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, πρέπει να μείνουν υπό έλεγχο οι εξελίξεις ε, αυτών των τελών ε, και να αποφύγουμε πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Καλό είναι να υπενθυμίσουμε από πλευρά Επιτροπή ότι οι οργανισμοί ρυθμίζουν διαφορετικού κλάδου και έτσι η θέσπιση τελών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Σημειώνουμε ε, τα συμπεράσματα και τα πορίσματα για την περιορισμένη δυνατότητα επέκτασης ε, του συστήματος τελών και των όσων αναφέρονται για την διερεύνηση εναλλακτική χρηματοδότησης όπως ε, η θέσπιση τελών με βάση την αξία. Πρέπει λοιπόν να τα διαρευνήσουμε όλα αυτά, αλλά πάντα έχοντας κατά νου και τις νομικές ε, συνέπειες για την Ένωση σε ό,τι αφορά την ίσπραξη τελών που ε, μοιάζουν με φόρους. Μια τελευταία παρατήρηση. Γι' αυτό που αναφέρεται στη μελέτη, ότι ε, πρέπει να αποφύγουμε μια μεγάλη, ένα άκαμπτο σύστημα. Υπάρχει μια τέτοια ακαμψία, αλλά θεωρούμε ότι αυτό ορθώς γίνεται. Γιατί οι δραστηριότητες ε, που βασίζονται ε, στα τέλη ε, έχουν μεταβαλλόμενο χαρακτήρα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ σημαντικοί στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οι ερευνητέ της Deloitte μας έδωσαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ECA που αναμένεται να μειώσει τα έσοδα από τα τέλη του μέσα στα επόμενα χρόνια και πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την πτώση σε σχέση με τον αριθμό του προσωπικού. Καθώς και τα αναμενόμενα έσοδα μπορούν να δημιουργήσουν την ανάγκη μεγαλύτερης ε, εξισορρόπησης μέσω επιδοτήσεων από τον ενωσιακό προπολογισμό. Τέλος, ενώ φαίνεται ότι είναι δωρεάν ουσιαστικά χωρίς περαιτέρω κόστος... για τον ενωσιακό προπολογισμό αυτές οι υπηρεσίες, εκ ε, μακροπρόθεσμα δεν ισχύει αυτό γιατί ε, ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός θα πρέπει να καλύψει το συνταξιδετικό πρόγραμμα αυτών των υπαλλήλων. Συνεχίζουμε λοιπόν να παρακολουθούμε με προσοχή την εξέλιξη τη θέσπιση τέτοιων συστημάτων στου οργανισμού. Υπενθυμίζω το πιλωτικό έργο τη ΕΑΖΑ, που είναι σημαντικό νέο στοιχείο από αυτή την άποψη. Ευχαριστώ και πάλι για την διοργάνωση αυτή τη ενδιαφέρουσα συζήτηση δώσουμε, θέλαμε να δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους ε, των ευρωπαϊκών οργανισμών. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά ε, μπορούν να μας στείλουν γραπτό στις παρατηρήσεις τους ε, και να μας πούν σε ποιο βαθμό θέλουν να προβλέψουν συμπληρωματικά τέλη. Γιατί όλα αυτά συνεπάγονται την μείωση του δημοσιονομικού αντικτύπου και αυξάνουν την ευελιξία του προπολογισμού μας. Φυσικά κάθε οργανισμός έχει ειδική προσταθεμένη αξία και ανταποκρίνεται στα κριτήρια αποδοτικότητας, ε, ανταγωνιστικότητας και αριστείας. Τώρα, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τιερή Σούμπρουκ για τρία λεπτά μόνο, γιατί ε, πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να απαντήσω μέσα σε τρία λεπτά όλα τα σχόλιά σας τα περισσότερα από αυτά τουλάχιστον, για τα πρώτα σχόλια ε, για την ενίσχυση της συνεργασίας και να είμαστε πιο προορατικοί σε ό,τι αφορά τον κλάδο. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε και από του οργανισμού, ότι πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κλάδο, πρέπει να υπάρξει ε, μια κοινή διαδικασία και αυτό βοηθάει. Ε, δεν έχουμε καταλήξει συμπέρασμα ότι υπάρχει προβληματική ε, πρόβλημα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας εξαιτία ε, του συστήματο επιβολή τελών. Κάποια σχόλια αφορούσαν τα ποσά, ότι τώρα είναι μόνο 34% και ότι οι δυνατότητε επέκταση είναι μόνο 3 με 4%. Με ρωτήσετε για, τα, για τους απόλυτους αριθμούς. Ουσιαστικά 90 έως 100 εκατομμύρια θα προκύψουν από αυτό το σύστημα. Ανάλογα με την ερμηνεία, η περιορισμένη αύξηση από το 34% στο 37% σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με τον χαρακτήρα των υπηρεσιών που βασίζονται σε τέλη, γιατί συνδέονται με διαδικασίες εποπτείας, ε, πιστοποίησης και για την πλειονότητα των οργανισμών δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα διασύνδεσης με τον κλάδο. Δεν έχουν λοιπόν αυτή τη δυνατότητα. Για την άλλη πηγή χρηματοδότησης, ε, τις ε, πληρωμές για, τις, ε, για την παροχή υπηρεσιών, εξηγήσαμε ότι είναι πολύ περιορισμένο το εύρος αυτών των δραστηριοτήτων, αυτών των υπηρεσιών και επίσης είναι περιορισμένη και η προβλεψιμότητα αυτών των υπηρεσιών. Γι' αυτό εκεί είναι μικρή η δυναμική τους για την αλλαγή του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεν προτείνει η μελέτη να μην υπάρξει κεντρική ε, εποπτεία των οργανισμών, ούτε ότι δεν πρέπει να υπάρξει απαλλαγή αυτών των οργανισμών. Απλώς ε, είπαμε ότι για λόγους εναρμόνισης αυτών των αρχών με βάση τα τέλη, καλό θα ήταν να απλουστευτεί το σύστημα. Άλλο ερώτημα αφορούσε την αναλογικότητα των τελών σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει κάποιο είδους ε, αναλογία με, ε, μεταξύ κόστους και υπηρεσίες. Δεν ισχύει πάντα αυτό, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αντικατοπτρίζει το τέλος το κόστος ε, που απαιτείται για την ε, παροχή της υπηρεσίας. Μετά, με ρωτήσατε για τους μικρότερους και μεγαλύτερους ε, φορείς και παίκτες, αν θέλετε, του κλάδους. Δεν ε, το εξετάσαμε στη μελέτη, αλλά λάβαμε υπόψη διαφορετικά ποσά τελών για μικρούς οργανισμούς, για να αποφύγουμε τις τρευλώσεις ε, της αγοράς προς τις μικρόμεσες επιχειρήσεις ή ένα ιδιαίτερο άκθος προς τους μικρούς οργανισμούς. Μετά, μιλήσατε για την κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ οργανισμών. Αυτό δυστυχώς ε, δεν ε, αποτελεί τμήμα της μελέτης μας. Δύσκολα θα μπορούσα να σχολιάσω κάτι τέτοιο. Άλλα σχόλια αφορούσαν τη δυνατότητα πιθανής εναρμόνισης τη συλλογή τελών από ό,τι κατάλαβα, γιατί όλοι αυτοί οι οργανισμοί έχουν διαφορετικά συστήματα συλλογή και ίσπραξη. φυσικά ο χαρακτήρας όλων αυτών των οργανισμών διαφέρει. Για παράδειγμα ο SRB που χρεώνει τέλη για ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Ε, διαφέρει κατάσταση σε σχέση με άλλους οργανισμούς που μπορεί να χρεώνουν διαφορετικά μέρη. Όπως και η μεθοδολογία υπολογισμού των τελών διαφέρει. Οπότε μπορεί να είναι δυνατή κάποια μορφή εναρμόνισης, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτά τα δύο στοιχεία που προανέφερα είναι σημαντικά και αποτελούν σημαντική διαφοροποίηση. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι τελειώνει ο χρόνος μου για το γλωσσάρι που αναφέρατε υπάρχει στην έκθεση στη σελίδα 6. Ελπίζω έτσι να σας βοήθησα και να μπορείτε πιο εύκολα να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, μάλλον ε, βιάστηκα ε, και σας πίεσα λίγο. Μπορείτε να μας στείλετε και γραπτό στα σχολιά σας ε, για όσους έρχονται τώρα. Ε, πρέπει να σας επαναλάβω ότι οι διερμηνείς βρίσκονται εδώ διότι είναι επιταγμένοι από τη διοίκηση ε, και γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε στις 10.30 ακριβώς γιατί δεν μας χορηγούν υπερβάσεις ωραρίου στο πλαίσιο της εργασιακής τους διάνοιξης με τη διοίκηση. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο. Παρακαλώ να βάλετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες ε, για δοκιμαστική ψηφοφορία στα μηχανήματα. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Για να δούμε, ψηφίσατε όλοι. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Πέραση ψηφοφορίας. Λοιπόν, για την εντολή, για τον τριμερή διάλογο καταρχάς. Κύριε Πρόεδρε, διακόπτη, μια βουλευτής, συγγνώμη δεν έχω την κάρτα μα. θα ψηφίζω δυνατάσω στις χειρός. Ωραία, το σημειώνουμε. Ωραία, μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία για την εντολή για τον τριμερή διάλογο 12 Ιουλίου για το σχέδιο προπολογισμού του 2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροπολογία 1, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε για την 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Il est repoussé. Απορρίπτεται. Τι ψηφίσατε κυρία Βαϊντέρε. Μάλιστα. Δεν μας ακούει. Απορρίπτεται ούτως ή άλλως. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Παρακαλώ, θα με βόλευε αν σηκώνατε και τα χέρια. Νομίζω απορρίφθηκε, αλλά θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 13. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 2 ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 ψήφι περ και 24. 23 και 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 ψήφι περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 26 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 27 ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται 28 ψήφι υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Γιατί αγαπητοί συνάδελφοι δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Για το 28 ξανά διανατάσεως υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε. 29 άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 29. Τροπολογία 30. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Να σηκώνετε τα χέρια. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Ισοψηφία. Κυρία Βέντερ όμως έχει ψηφίσει κατά, άρα απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 έχει αποσυρθεί. 36 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 ψήφι Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 44 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 60 ψήφι υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την 60 άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 14 προς 11 61 ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 ψήφι περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 ψήφι περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 με προφορική από τον εισηγητή περ. κατά, αποχές εγκρίνεται. 66 ψήφι κατά, αποχές απορρίπτεται. 67 με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 70 έχει αποσυρθεί. 71 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την 72 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία συγκρίνεται 13 προς 11. Κύριε Βάιντερ, εσείς σας φέραν την κάρτα, ωραία. Η επόμενη με προφορική, η παράγραφος 23 δηλαδή, εγκρίνεται 73 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 75, 74 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108 υπέρ, α, συγγνώμη, έχει καταπέσει. 108 έχει καταπέσει, πράγματι. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία έμπλ 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κάλτ 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Φαμ 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε. Ορίστε. Θέλετε. Δεν το ψηφίσαμε το ΦΑΜ 1. Α, θέλετε έλεγχο. Μάλιστα. Θέλετε έλεγχο για την τροπολογία ΦΑΜ 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε 14 ή 15 προς 2. Προς 12, συγγνώμη. Απορρίφθηκε. Για το σύνολο του κειμένου, ονομαστικά ψηφίζουμε, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι? Όχι. Ένας από σας δεν έχει ψηφίσει. Δεν θα περιμένουμε όμως επαόριστον, οπότε πέρασε ψηφοφορία. 20 υπέρ, 4 κατά, μία αποχή. Εσεί, κυρία Βαϊντέρε. Α, ναι, με συγχωρείτε, έχετε την κάρτα σα, το ξέχασα. Ωραία. Naturellement, je félicite notre rapporteur. Να συγχαρούμε τον εισηγητή, τον κύριο Κλωτή. Με τέτοια ψηφοφορία δεν θα δυσκολευτούμε να μας ακούσει, να ακούσει τις απόψεις μας στο Συμβούλιο. Πολλά υποσχόμενο το γεγονός τώρα. Θα δούμε το σχέδιο τροποποιητικού προϋπολογισμού 2018 που κατά βάση σχετίζεται με την διευκόλυνση που παρέχεται στην Τουρκία για την υποδοχή ε, προσφύγων και μεταναστών από τη Συρία. Αν δεν έχετε πρόβλημα θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε αν μπλοκ τις 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Όχι. Λοιπόν, 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Scrutin est clos. Repoussé par 14 voix contre 12. 14 εναντί 12, 3 υπέρ, κατά. αποχέ, απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά. αποχέ, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά. απόχέ, απορρίπτεται. Ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία εγκρίνεται 20 υπέρ 4 20 Τέσσερις κατά δύο αποχές. Ε, ο Γενικός Συγητής, τον οποίο δίνω το λόγο σε σχέση με τις ε, τροποποίησεις των μεταφορών πιστώσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέντε με... αιτήματα μεταφορών πιστώσεων πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα το πρωί για το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας ε, για παροχή βοήθειας σε πολλές χώρες ε, που επλέγησαν από φυσικές καταστροφές ε, και από εκτοπισμούς πληθυσμών. Μιλάμε για συνολικά 120 εκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. Θα μιλήσω για όλες μαζί κύριε Πρόεδρε, διότι δεν δημιουργούν πρόβλημα και προτείνω να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Η πρώτη πρόταση είναι η απόφαση 12 της Επιτροπής αφορά την Αιθιοπία όπου εκτιμάται ότι 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά από το Μάιο του 2018 λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 35 εκατομμύρια προτείνω να μεταφερθούν από το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης για την παροχή ανθρωπιστικής αρρωγής στους εσωτερικά εκτοπισμένους πληθυσμούς οι οποίοι δεν λαμβάνουν από αλλού καμία υποστήριξη. Θα εστιαστούμε στην επίγουσα στέγαση, διατροφή και στην παροχή των βασικών για τη διαβίωση, για νερό, για έκτακτες ανάγκες και για παιδεία. Προτείνω να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτό για την Αιθιοπία. Μετά έχουμε την απόφαση 13 αφορά το Κόγκο, όπου είχαμε ε, τον ιό έμπολα, πάλι κρούσματα ε, και την κλιμακούμενη βία. 35, 25 εκατομμύρια ευρώ προς τους ε, πληθυσμούς αυτούς που επλέγησαν από τον έμπολα, από που έπεσαν θύματα παρακολούθησης και βίας. Η τρίτη μεταφορά είναι το Σουδάν. όπου οι άνθρωποι που χρειαζόνται ανθρωπιστική βοήθεια αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατομμύρια τους τελευταίους μήνες. Γι' αυτό το λόγο διαθέτουμε 10 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της επιδεινούμενης κατάστασης, κατάστασης ασφαλείας. Τα χρήματα θα πάνε εκεί επίσης για σωστή διατροφή αυτών των ανθρώπων. Η απόφαση 15 αφορά το Τσάντ, το Καμερούν και την Ιγυρία και εκεί έχουμε εκτοπισμένου πληθυσμού 30 εκατομμύρια ευρώ. Επίση για βοήθεια διατροφή και για διατροφή επιβίωση για ανθρώπου που βρίσκονται σε δινή κατάσταση. Και απόφαση 16 Αφγανιστάν 20 εκατομμύρια λόγω τη ε, ξηρασία ε, που υπάρχει εκεί. Δεν χιόνισε αρκετά το χειμώνα στο Αφγανιστάν. Γι' αυτό δεν υπάρχει αρκετό νερό. Η γενική κατάσταση ασφαλείας επίσης ε, είναι δύσκολη. Για αυτό το λόγο διαθέτουμε 20 εκατομμύρια ευρώ για την παροχή πιο συγκεκριμένα νερού, αλλά και για να βοηθήσουμε τους εσωτερικά εκτοπισμένους πληθυσμούς και τους ανθρώπους που επλήγησαν από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. καθώς επίσης και επειδή το Αφγανιστάν αναμένει την επιστροφή ενός εκατομμυρίου ανθρώπων από το Ιράν και το Πακιστάν φέτος. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται περαιτέρω υποστήριξη. Πέντε αποφάσει λοιπόν για ανθρώπου που χρήζουν βοήθεια σε αφρικανικέ χώρε και στο Αφγανιστάν. Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να τα ψηφίσουμε όλα μαζί, όλε αυτέ τα αιτήματα και να τα ψηφίσουμε υπέρ. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Εισηγητά. Υπάρχουν ερωτήσει ή παρατηρήσει. Δεν βλέπω. Α, Λοιπόν, ο Γενικό Συγητή μα καλεί να ψηφίσουμε unblock και τι πέντε αυτέ μεταφορέ πιστώσεων. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, συγγνώμη. Θα ξανακάνουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ε, 24 υπέρ, μία κατά, δύο αποχές. Το λόγο έχει ο κύριος ε, Ashworth που θα μας προτείνει μεταφορές ε, σε επίπεδο ε, Επιτροπής Περιφερειών που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. ήθελε συμπληρωματικές πληροφορίες ο κύριος Ashworth, μεταφορές για την ΕΟΚΕ, ελεκτικό συνέδριο και Επιτροπή των Περιφερειών, δυνάμει του άρθρου 25 του Οικονομικού Κανονισμού. Έχετε το λόγο, κύριε Ashworth. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω είπατε, έχω διάφορε μεταφορέ πιστώσεων αυτή την εβδομάδα. Καμία δεν δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα και καμία δεν απαιτεί ψήφο. Θα σα τι ε, περιγράψω όλε. Όπω είπατε, η πρώτη αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών. Μεταφορά 60.000 ευρώ για νέα συστήματα πληροφοριών στο κτίριο Ζακτελόρ. Θα θυμάστε ότι αυτό αναβλήθηκε από την περασμένη εβδομάδα γιατί δεν ήθελα να κάνω περαιτέρω ερωτήσει. Ε, είμαι ικανοποιημένο από την απάντηση που έλαβα ότι οι οικονομίες ε, θα βρεθούν ε, από τις αποζημιώσει λόγω του χαμηλότερου από τον αναμενόμενο προπολογισμό στο Βέλγιο φέτος. συγγνώμη για την ΕΟΚΕ 175.000 ε, ευρώ για, την, ε, για οθόνες στο κτίριο Ζαγντελόρ αλλά και για τεχνικό εξοπλισμό αντικατάστασης παλιού εξοπλισμού σε διάφορες αίθουσες συνεδριάσεων. Δεν απαιτείται ε, ψηφοφορία. Ωστόσο δύο σχόλια έχω να κάνω. Πρώτον, εγκρίνω την έγκριση του εξοπλισμού αυτού, ένα κομμάτι του οποίου ήταν φορητά ε, συστήματα ε, ψηφοφορίας για τις συνόδους ε, της ΟΚΕ που λαμβάνουν χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ νομίζω ότι το δικό μας σύστημα ήταν επαρκές. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Επίσης αλλά ένα σχόλιο όταν συντάσσουμε τον προπολογισμό. Η μετάφραση, το κόστος μετάφρασης ήταν μη διαπραγματεύσιο με την ΕΚΟΣΟΚ μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει περιθώριο ελιγμών. Αλλά τώρα ξαφνικά βρήκαμε οικονομία 175.000 ευρώ από τη μετάφραση. Απλά το σχολιάζω με κάποια έκπληξη. Τρίτο σημείο αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Επτά αιτήματα μεταφοράς πιστώσεων έχουν. Δεν θα τις δούμε όλες λεπτομερώς. Είναι μικρά ποσά. τα σχέδια έχουν λάβει ερωτήσει. Ε, ε, το ελεκτικό συνέδριο έχει διαπιστώσει διάφορε εξοικονομήσει σε διάφορε αποζημιώσει και θα χρηματοδοτήσει νέο φόρτο εργασιών ε, και το κόστος μετάφραση όταν αντίθεται σε τρίτου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα αίτημα απελευθέρωση κονδυλίων, αποδέσμευση κονδυλίων για οκτώ ε, συμβασιούχους που θα αναλάβουν το φόρτο εργασίας που σχετίζεται με τους Βρετανούς μέλη του Κοινοβουλίου και επιπλέον συμβασιούχοι που θα αρχίσουν να δουλεύουν στο Ευρωπαϊκό Κόμβο ε, Μέσων και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ε, ζήτησε 76.000 ευρώ για περαιτέρω χρηματοδότηση εκπαιδευόμενων ε, και μετάφραση λόγω των αυξανόμενων δραστηριοτήτων ε, του τμήματος της ε, Διαμεσολαβήτριας. Όπως είπα, δεν απαιτείται ψηφοφορία. Συνιστώ να εγκρίνουμε όλα αυτά τα αιτήματα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σιγητά. Σημειώσαμε τη θετική σας ε, γνώμη για όλες αυτές τις μεταφορές. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, θεωρώ ότι εγκρίνονται. Α, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω ψηφοφορία για μία από τις ε, μεταφορές πιστώσεων σε ό,τι αφορά το αίτημα του ελεγκτικού συνεδρίου για 516.000 ευρώ. ecavabo 4 t 18 συγκεκριμένα, Αναφέρεται στην αιτιολόγηση ότι θέλουν να αξιοποιήσουν 150.000 από αυτό το ποσό για να δώσουν ηλεκτρονικές ε, ταμπλέτες στα μεσαία στελέχη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι σωστή αξιοποίηση των χρημάτων φορολογουμένων. Και για να σας δώσω ένα ακόμα τέτοιο παράδειγμα κακής, ε, κακού προγραμματισμού δημοσιονομικού, εφόσον έχουμε δει και πολλές ε, από αυτές ε, τις αιτήσει για μεταφορά πιστώσεων και πολλές από αυτές δεν είναι και ορθώς αιτιολογημένε. Εντάξει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς είμαστε κατά ε, της υπέρβασης των πιστώσεων σε ό,τι αφορά το ελεγκτικό συνέδριο. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό είμαστε υπέρ κάθε μεταφοράς επίστοσης ε, για το ελεγκτικό συνέδριο. Αλλά για τα, όλα τα υπόλοιπα να θεωρήσετε ότι τα καταψηφίζουμε. Ωραία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Α, ποιος άλλος θέλει το λόγο. Oui, vous en prie, vous avez la parole. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ, πλευρά μου, θα ήθελα να πω ότι, σαν πολιτική ομάδα, είμαστε υπέρ τη πρόταση του εισηγητή, αλλά επί τη ευκαιρία να τον συγχαρώ για όλη τη δουλειά που έχει κάνει, γιατί τις περασμένες εβδομάδες ε, κατάφερε να συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες που είναι σημαντικές παρά τις αμφιβολίες μας. Ε, γι' αυτό τον λόγο τον ε, στηρίζω ε, στη μεταφορά πιστώσεων. Τώρα για το ελεγκτικό συνέδριο έγινε μια παρατήρηση, αλλά πρέπει να επισημάνω ότι δεν πρόκειται για το μόνιμο προσωπικό Πρόκειται για προσωπικό που κινείται εκτός του ελεγκτικού συνεδρίου. Γι' αυτό και χρειάζεται ε, αυτά τα τάμπλετ. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο? Όχι. Συνάδελφοι, προτείνω να θεωρήσουμε ότι ε, εγκρίνονται οι δύο μεταφορές πιστώσεων για τις οποίες δεν υπάρχει επιφύλαξη και μετά ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε για αυτή την, ε, τη ΣΕ 18 για το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, οπότε άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Σκοτάει κλού. Πέρασε. Εγκρίνεται. 26 ψήφοι υπέρ, συγγνώμη, 23 υπέρ, 3 κατά, 0 αποχές. Η Μόνικα Χολμάγερ τώρα να μας παρουσιάσει σύντομα το φάκελο που ήδη έχει συζητηθεί και κλεισμένο το θηρόν την περασμένη φορά, στην περασμένη μας συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, από τη διοίκηση βλέπουμε ότι έχουν δοθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα στους σκιώδεις εισηγητές. Κάναμε λοιπόν ε, μια συζήτηση στο μέλλον. Ελπίζω βέβαια τα έγγραφα να παρέχονται στον εισηγητή και στους σκιώδεις ε, εκ των προτέρων για να υπάρχει ο απαραίτητο χρόνο να τα εξετάζουμε. Και εμεί θα διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν εμπιστευτικέ πληροφορίε, όπω για παράδειγμα ε, τα κεφάλαια για κονδύλια που συνδέονται με, τα security, με, συγγνώμη, ζητήματα ασφάλειας, τα οποία μπορούν να κρυπτογραφηθούν ε, και έτσι να δοθούν στα μέλη της Επιτροπής. Συμφωνούμε κατά λοιπά ότι είναι εμπιστευτικός ο φάκελος, γιατί είναι ευαίσθητο ζήτημα ως προς την ασφάλεια. Προφανώς και δεν γίνεται να δημοσιοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία αν θέλουμε να μεριμνήσουμε για την ασφάλεια. Για το κτίριο Λουίς Βάης τώρα. Πρώτα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος ελέγχου ασφαλείας που δεν βρίσκεται τη στιγμή εντός ε, του Κοινοβουλίου. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Να υπάρχει ένα ξεχωριστό κέντρο πιστοποίησης για τους επισκέπτες. Να μην είναι εντός του κτιρίου, δηλαδή και πάλι. Να γίνεται αυτή η πιστοποίηση πριν μπει κάποιο στο κτίριο. Και να έχουμε καταστάσεις και για τις ε, ομάδες ε, και που επισκέπτονται το κοινοβούλιο και για τους μεμονωμένους επισκέπτες, το οποίο είναι το πρόβλημα μέχρι σήμερα. Είναι μικρό το κτίριο. Δεν χωράνε πολλοί άνθρωποι μέσα ταυτόχρονα. Ενώ συνήθω έχουμε πολύ περισσότερους επισκέπτες κάθε μέρα ε, στο Στρασβούργο. 1.700 τετραγωνικά μέτρα, περίπου 25 μήνες ε, μέχρι να ε, κατασκευαστή. Τώρα, τις πληροφορίες σας τις έχουμε δώσει. Ζητώ λοιπόν την έγκρισή σας, Πρόεδρε. Bien, merci. Ωραία, ευχαριστούμε την κυρία Συγήτρια. Δεν ζητάει κανείς το λόγο. Θα ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 ψήφοι υπέρ, μία κατά, τρεις αποχές. Σε στην εισηγητρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω απλά ότι στο πλαίσιο του δημοσιο... πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου το συζητάμε αυτό για τη μία έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν γίνει διάφορες δηλώσεις από τη Γαλλία για τη Γερμανία ότι η μία έδρα συμφέρει και την Προεδρία. Οπότε νομίζω είναι σαφές ότι η συνθήκη της Λισαβόνας ε, αναφέρει φυσικά το Στρασβούργο ως έδρα, οπότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να βεβαιωθούμε ότι η έδρα θα είναι το Στρασβούργο και έτσι θα συνεχίσει και στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα κόστη και να ζητήσουμε τις υπηρεσίες μας να μας δώσουν κάποιες επιλογές στρατηγικές για το τι θα σημαίνει όλο αυτό. Ε, αν είναι να φύγουμε από τις Βρυξέλλες και να πάμε στο Στρασβούργο το οποίο θα έχουμε ορίσει ως ενιαία έδρα του Κοινοβουλίου. Κύριε Ρούμπικ, ε, πολύ προσωπικά εγώ δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που προτείνεται, αλλά δεδομένης της ώρας ε, που έχει πάει και των περιορισμών και ότι πρέπει να σταματήσουμε την ψηφοφορία πριν τις 10.30, θα αναβάλουμε και αργότερα τη συζήτηση αυτή. Αλλά παρατηρούμε ε, τις, τις παρατηρήσεις τι σημειώνουμε. Θα ψηφίσουμε τώρα επί του ψηφίσματος για την ε, παράταση της λίστας χωρών Σε οποίες μπορεί να δανείσει η ε, ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Παράταση λοιπόν για το Ιράν. Έχει γίνει έτοιμα ξεχωριστής ψηφοφορίας σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Θα το δούμε ηλεκτρονικά. Πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 21 εναντί 4, ε, 2 υποπρόεδρος αλλά είναι 4. Δεύτερο τμήμα. και καταπίπτει και τώρα πάμε να ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου έτσι όπως δεν τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, όχι συγγνώμη, απορρίπτεται 22 έναντι 4. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν τις ψηφοφορίες. για την πολιτική ακινήτων που άρχισε να αναφέρει ο κύριος Ρούμπικ. Ε, κυρία εισηγήτρια, έχετε να κάνετε κάποια ανακοίνωση. Όχι. Ωραία, λοιπόν, να σας ζητήσω αγαπητοί συνάδελφοι, αν έχετε κάτι να συζητήσουμε από τα διάφορα. Όχι. Κύριε Ντεμπρέ. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να μάθω γιατί αλλάξαμε τη θέση της ομάδας μου ε, Εντό τη συνεδριάσεώ μα. Εδώ και τέσσερα χρόνια είμαστε από τη μια πλευρά και για πρώτη φορά βρέθηκα σε αυτή την πλευρά εδώ. Γιατί μας άλλαξαν τη θέση. Με ποιο κανόνα έγινε αυτό. Μα προάγεται ή μας τιμωρείται ή έγινε κάποιο σφάλμα. Αυτό που αισθάνεστε θα πρέπει να το αισθάνεται ο καθένα μα, ξέρετε. Ο μόνο που δεν μετακινήθηκε είναι ο πρόεδρο. Ωραία. Δεν υπάρχουν ε, θέματα υπό τα διάφορα. Η επόμενη συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφοι, στο Στρασβούργο, που μπορεί να γίνει η έδρα, που εξακολουθεί να είναι η έδρα, όπω είπε και ο κ. Ρούμπεξ, σας το επιβεβαιώνω, δυνάμει των συνθήκων, 2 Ιουλίου, Δευτέρα, με την ΕΚΟΝ. Νομίζω ότι είναι στις 7.30, όχι, στις 8.45 ε, το βράδυ, 9 παρατέταρτο το βράδυ. Δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Πέρα τη σα.